χρόνια και η Προεδρία μας θα εξασφαλίσει ότι παραμένει το θέμα αυτό στην ατζέντα μας. Σε ό,τι αφορά το πώς θα αντιμετωπίσουμε τη διαδικασία του άρθρου 7 στην Πολωνία, πώς θα την αντιμετωπίσει το Συμβούλιο, ξέρετε ότι η Προεδρία δεν μπορεί να προδικάσει τις συζητήσεις του Συμβουλίου και να προβλέψει και το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων. Όλε οι πρόσφατε νομοθετικέ εξελίξει στην Πολωνία τι παρακολουθούμε, ούτω ώστε το Συμβούλιο να έχει μια πλήρη εικόνα για την κατάσταση και να έχουμε τα θεμέλια για να πάρουμε τις μελλοντικές μας αποφάσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ένα ψήφισμα υποβλήθηκε από πέντε πολιτικές ομάδες σχετικά με τις ακροάσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 σχετικά με την Πολωνία και την Ουγγαρία. Έκλεισε η συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί αύριο. Και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης την δήλωσή του Συμβουλίου και της Επιτροπής σε σχετικά με την επανάληψη της ποινική διαδικασίας κατά του Πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας για κατάχρηση κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Κυρία Βρενιάτ, σας, σας δίνω πάλι το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ ξανά. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας διαβεβαιώ το Συμβούλιο δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο να εξασφαλίσει ότι τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούνται με βάση τους κανόνες και σέβονται τις αργές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Γνωρίζω τους ισχυρισμούς στα ΜΜΕ εναντίον του Τσέχου Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, σε ό,τι αφορά την, ε, τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ε, Ευρωπαϊκών Διαρθωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Οι τσεχικές αρχές διερευνούν την υπόθεση. Ξέρετε ότι δεν μπορεί το Συμβούλιο να σχολιάσει τις εθνικές αυτές ε, διαδικασίες που είναι εξελίξη. Θα ήθελα να τονίσω εδώ ότι είναι σημαντικό να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει σωστά το έργο της. Επίσης γνωρίζω ότι η Κομισιόν, όπως είπε στην Ολομέλη του Δεκεμβρίου, έχει κάνει έναν έλεγχο και θα ακούσω τι θα μας πει η Κομισιόν σήμερα. Σας διαβεβαιώ ότι συμφωνούμε ότι είναι υψής της σημασίας ε, να υπάρχουν ισχυροί μηχανισμοί για να προστατευτούν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και να εξασφαλίσουμε ότι τα λεφτά ξοδεύονται με κατάλληλο και ένομο τρόπο. Το Συμβούλιο είναι υπέρ διαφόρων πρωτοβουλειών για να προστατεύσουμε ακόμα περισσότερο τα δημοσιονομικά και οικονομικά συμφέροντα τη Ένωση. Παραδείγματο χάρη, ε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα αρχίσει να λειτουργεί φέτο το 2020 ή την οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης αντίον των, ε, οικονομικών σφαιρών της Ένωσης με την ποινικοποίηση τέτοιων ε, τάσεων. Θα ακούσω πολύ προσεκτικά λοιπόν τη συζήτησή, μα, τη συζήτησή σας. Ευχαριστώ. Danke. Σας ευχαριστώ. Επιτρόπος Σινκεβίτσιους έχει το λόγο τώρα. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει την κατάσταση στο θέμα αυτό. Τρία πράγματα θα ήθελα να καταστήσω σαφή από την αρχή. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μηδενική ανοχή σε περιπτώσεις κατάχρησης κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, πάντα ε, δίνει συνέχεια σε ε, αναφορές ε, σύγκρουσης συμφερόντων σε όλα τα κράτη-μέλη. Τρίτον, ε, έχει αναλάβει ευρεία και στονισμένη δράση όσον αφορά ε, τις φερόμενες συγκρούσεις συμφερόντων ε, στην Τσεχική Δημοκρατία. Ποια είναι τα γεγονότα και πού βρισκόμαστε στη διαδικασία ελέγχου. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής έκαναν ελέγχους τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2019 στην Τσεχική Δημοκρατία οι οποίες σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο για την Ανάπτυξη της Υπέθρου. Ε, σε διαφορετικά στάδια της διαδικασίας βρισκόμαστε όσον αφορά τα διάφορα αυτά ταμεία. Για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, ε, βρίσκονται τώρα πια στο τελικό στάδιο ενώ η έκθεση που έχει δοθεί στην Τσεχία δεν αποτελεί την τελική φάση της διαδικασίας. Το περιεχόμενο της τελικής έκθεσης θα παραμείνει εμπιστευτικό μέχρι το κλείσιμο της διαδικασίας, δηλαδή μέχρι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει ε, λάβει οριστική θέση. όσον αφορά τη, τα μέτρα επένδυσης για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει επιστολή στο κράτος μέλος αυτό με, κάποιες κάποια πρώτα συμπεράσματα και συστάσεις για την αποφυγή σύγκρουση συμφερόντων στο μέλλον. Η διαδικασία συνεχίζεται και το επόμενο βήμα θα είναι διμερή σε συνάντηση με τις τσεχικές αρχές. Για όλα τα ταμεία η διαδικασία μέχρι την πιθανή επιβολή διορθωτικών ε, μέτρων ε, μπορεί να διαρκέσει μέχρι 20 μήνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει μια δίκαιη διαδικασία. Ο πρώην Επίτροπος Ότινγκερ και τώρα ο Επίτροπος Χάν έχουν ε, στείλει σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και κλεισμένων των θυρών. Δεν θα σχολιάσω σήμερα τα συμπεράσματα λόγω εμπιστευτικότητα. Όσο συνεχίζονται οι έλεγχοι, ο προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση προστατεύεται απολύτω. Δεν γίνονται πληρωμέ από τα ταμεία αυτά σε προγράμματα όπου μπορεί να υπάρχει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά το Ταμείο Ανάπτυξης της Υπέθρου. Δεν επιστρέφονται δαπάνες ε, στην Τσεχία για έργα όπου πιθανότατα να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Να πω τώρα λίγα λόγια ε, για για την ε, φωλιά του πελαργού δόθηκε χρηματοδότηση το Δεκέμβριο του 2017. Ο Όλαφ ολοκλήρωσε τις έρευνές του και ε, συνέστησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακτήσει το σύνολο της επιδότησης. Επίσης, ε, συστήθηκε στις ε, αρμόδιες αρχές της Τσεχίας να λάβει υπόψη τα συμπεράσματα ε, του Όλαφ. Οι τσεχικές αρχές απέσυραν από την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση το έργο αυτό και ανέκτησαν τις επιδοτήσεις από τον δικαιούχο. ενώ η συνέχιση τη έρευνα αυτή είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των σεχικών τέλο. Τέλος, όσον αφορά ε, άλλα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης ε, θα εξετάσει περιπτώσεις ε, συγκρούσει συμφερόντων σε άλλα κράτη-μέλη. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει στήριξη σε όλα τα κράτη-μέλη για να εφαρμόζουν σωστά μέτρα σε περιπτώσει σύγκρουση συμφερόντων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σεντεχόφσκι έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Ε, κύριε εκπρόσωπε του Συμβουλίου, ενώ η συζήτηση αυτή έχει να κάνει με ε, λογιστικούς ελέγχους και έρευνες, ε, ας προχωρήσουμε σε πιο γενικό επίπεδο. Ας εξετάσουμε ποιες είναι οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επανειλημμένα, ο Επίτροπος Χαχάν μας διαβεβαίωσε ότι ισχύουν οι ίσες συνθήκες ανταγωνισμού για όλους. Ε, θα σας πω όμως τι συμβαίνει στην Τσεχία όταν υπάρχει ε, κάποιο λάθος ε, σε περίπτωση που αφορά ε, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Αμέσως γίνεται έλεγχος, αμέσως ε, γίνεται αίτηση ανάκτησης ε, επιστροφής των χρημάτων και αμέσως μόλις παραβιαστεί το δίκαιο της Τσεχίας ξεκινάει μια έρευνα. Αυτό όμως δεν συνέβη αυτή τη φορά. Έχουμε νέο κανονισμό και ο Πρωθυπουργό ε, συμμετείχε στην εκπόνηση του κανονισμού αυτού ως ε, Υπουργό ε, Οικονομικών. Και τώρα που ισχύει γι' αυτόν αυτός ο νέος κανονισμός δεν μπορούμε να τον εφαρμόσουμε. Το Συμβούλιο είπε ότι δεν θα επέμβει στις ε, τρέχουσες ε, έρευνες. Το ε, δεχόμαστε αυτό, αλλά θέλουμε σαφή δήλωση. Πρωθυπουργός που σύμφωνα με την λογιστική έκθεση είναι συνυπεύθυνος για θέματα προϋπολογισμού, εάν επιτρέπεται να κάνει τέτοια πράγματα. 1,5 λεπτό έπρεπε να μου έχετε δώσει. Δεν ξέρω αν πράγματι έχει λήξει ο χρόνος μου. Βόλτερς, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το Νοέμβριο 200.000 άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά του Πρωθυπουργού Μπάμπη στην πράγμα Και μετά ο κύριος Μπάμπης ε, επέμενε ότι η διαδήλωση και η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν μέρη, ε, μέρος μιας ε, προσπάθειας υπονόμευσης της εξουσίας του και αντιδημοκρατικές κινήσει. Είναι θεωρία συνωμοσία αυτό. Αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι νόμιμο καθήκον τη. Και επίση είναι καθήκον τη ε, απέναντι στου Τσέχου πολίτε που ζητούν δικαιοσύνη. Η ε, έκθεση τη Ελεκτική Επιτροπή, τη Επιτροπή που διέρευσε, ε, δείχνει ότι υπήρχε σαφή σύγκρουση συμφερόντων στην περίπτωση του κ. Μπάμπη, επειδή υπεξαίρεσε χρήματα των φορολογουμένων για προσωπικό του όφυλο. Τα εκατομμύρια που συζητιούνται εδώ πρέπει να επιστραφούν και χρειάζεται ο μηχανισμό κράτου που έχει προταθεί να εφαρμοστεί για να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία των ε, θεσμικών οργάνων επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Α βοηθήσουμε του Τσέχου πολίτε σήμερα και α αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει τη δουλειά τη. Ευχαριστούμε. Η Αντιπρόεδρος Χαραντσόβα. Μικρόφωνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Αρκετοί από εσά με γνωρίζετε καλά και οι περισσότεροι συνάδελφοι γνωρίζουν ότι ποτέ δεν ε, είχα αντίρρηση για μια επικοδομητική συζήτηση για οποιοδήποτε θέμα. Όμω θα πρέπει μια επικοδομητική συζήτηση να βασίζεται και σε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία και αυτό δεν ισχύει σήμερα. Ε, μιλάμε για εντυπώσει προσωπικέ έχθε κάποιε φορέ για την άποψη του καθενό. Ε, και έχει φτάσει αυτό να γίνεται συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ε, έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Ελεγκτική Επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η όλη αυτή η δικασία αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Δημοκρατία τη Τσεχία. Σε όλα τα υπόλοιπα, οι αρχέ τη χώρα, τη Τσεχία, κάνουν αυτό που είναι το καθήκον του και από νομική ε, σκοπιά η δικαιοσύνη στη χώρα εργάζεται όπω ε, θα έπρεπε, χωρί να παρακολείται από κανέναν. Οι διαδικασίε αυτέ θα εξακολουθήσουν ασχέτω τη συζήτηση εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι η συζήτησή μας είναι άσκοπη και δεν ε, έχει και λόγο ύπαρξης. Πρέπει λοιπόν να το δηλώσω. Η συζήτηση αυτή είναι, εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες και είναι μια ακόμη από τις προσπάθειες ε, κάποιων τσέχων συναδέλφων να επηρεάσουν τα πράγματα. Στην πραγματικότητα το Ευρωκοινοβούλιο έχει παρασυρθεί σε μια συζήτηση για τα εσωτερικά πολιτικά πράγματα της Τσεχίας και αυτό είναι απαράδεκτο και πλήττει την αξιοπιστία μας ως Ένωσης. Ευχαριστούμε. Η κυρία Φων Κραμών τον Παντέλ. Έχει το Πρόεδρε, συνάδελφοι, η κατάσταση στη δημοκρατία της Τσεχίας μας ανησυχεί. Ένα από του πλουσιότερου ανθρώπου στην Τσεχία, ο κ. Μπάμπη, αποφασίζει για τα πολιτικά πράγματα τη χώρα και ταυτόχρονα ψηφίζει και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την πολιτική συνοχή και τι διευθυντικέ πολιτικέ που τον έχουν κάνει πλούσιο. Εδώ μιλάμε για πραγματική σύγκρουση συμφερόντων. Όμω δεν θα πρέπει να αυταπατώμεθα. Εδώ δεν είναι το, η πηγή του προβλήματο ο κ. Μπάμπη, είναι ένα από τα συμπτώματα. Ε, όπου βλέπουμε αν υπάρχουν τέτοια προβλήματα στη χώρα, έχει παντού σχέση εκείνο με τα μέσα μαζική ενημέρωση, με τομέα τη οικονομίας και θα πρέπει να δούμε τα οικονομικά συμφέροντα, πώ έχουν διαπλακεί και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Η Σλοβακία και πολλέ φορέ και η Γερμανία. Ε, εδώ λοιπόν μιλάμε για έναν από πολλού ολιγάρχε που υπάρχουν αυτή τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν γίνει πλούσιοι με ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό που πραγματικά μα σοκάρει είναι ότι δεν ξέρουμε σε τι ε, διαστάσει ε, είναι ο κύριο Μπάμπη, εκείνο που έχει υποφεληθεί περισσότερο από όλου από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έχουν πολλέ πληροφορίε και θα μπορούσαν να ερευνήσουν περαιτέρω πού ακριβώς πηγαίνουν τα κονδύλια των διαφορετικών ταμείων τη της ε, κοινή αγροτική πολιτική. Χρειάζεται ε, κατεπηγόντω περισσότερη διαφάνεια. Χρειάζεται ένα σύστημα για να εντοπίσουμε αυτέ τι ατασταλίε, ε, τι παραβιάσει του συστήματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρί καθαρού κανόνε για την καταπολέμηση τη έκρουση συμφερόντων, χωρί καθαρού κανόνε για να ε, βρίσκουμε αυτέ τι παράνομε συμπεριφορέ, να τι διαλευκάνουμε, δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα. Χωρί όμω πολιτική πίεση για, τις, για τα ιστορικά πράγματα μια χώρα χώρα, την ιδιοκτησία των ανθρώπων αυτών. Τότε θα επιληθεί το θέμα αυτό, όταν ο εκδημοκρατισμό μετά το τέλο του κομμουνιστικού καθεστώτο επιτρέψει, ε, επιτρέψει στα κράτη που ε, βρίσκονταν ε, προηγουμένω στο κομμουνιστικό καθεστώ να κάνουν πραγματική πρόοδο. Το αγροτικό σύστημα άλλαξε τελείω, ιδιωτοποιήθηκαν τα πράγματα και αυτό βεβαίω ωφέλησε κάποιε πολιτικέ ελίτ. Κανόνε υπάρχουν. Αυτό ισχύει. Θα πρέπει λοιπόν η κρατική ιδιοκτησία να ενισχυθεί μεν, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην χειροτερεύει τα πράγματα δίνοντα τι μεγάλε πληρωμέ στου μεγάλου γεωκτήμονε στι χώρε αυτέ και όχι σε εκείνου που πραγματικά ασχολούνται με τι αγροτικέ δραστηριότητε και θα έπρεπε να ενισχύονται με τι επιδοτήσει. Ευχαριστούμε ο κύριος Ντάβιτ. Eh, Δεν είμαι φίλος eh, του Πρωθυπουργού Μπάμπης και διασώτης του. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η δημοκρατία. Αυτό σπούδασε σε, σε μια προνομιακή σχολή, μετά μπήκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα, στη μυστικές υπηρεσίες, εκπροσώπησε την Τσεχία στο εξωτερικό, στο κομμουνιστικό καθεστώς και μετά το 89, κατά τη διάρκεια των ιδιωτικοποίησεων, άρπαξε, υπεξαίρεσε, φετερίστηκε. Ε, βιομηχανικές παραγωγικές μονάδες στην παραγωγή τροφίμων και στη γεωργία και στα ΜΜΕ. Και επειδή ήταν πολύ καλό στο μάρκετινγκ, και επειδή οι ανταγωνιστές δεν ήταν τόσο καλοί όσο αυτός, κατάφερε να προωθήσει και το πολιτικό του project. Και το 2013 δίστησε στο Κοινοβούλιο και συνεχεία στην κυβέρνηση. Ε, συνεχεία κέρδισε τις γενικές εκλογές, τις βουλευτικές εκλογές και έγινε πρωθυπουργό. Οι εταιρείε του λαμβάνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία σε μεγάλη κλίμακα. Και η αντιπολίτευση τον ανάγκασε όμως να βάλει τις εταιρείε αυτές σε καταπιστεύματα. Στην πραγματικότητα εποφελείται μέσω των εταιριών του. Δημιούργησε άλλες εταιρείες στον τομέα της ψυχαγωγίας και το δικαστήριο θα αποφασίσει τι θα γίνει με αυτή την ε, επιχείρηση. Σε ό,τι αφορά τις διαδηλώσεις που τις ε, υποστηρίζει η αντιπολίτευση, κοστίζουν πολλά λεφτά. Αλλά οι προτιμήσεις του Πρωθυπουργού έχουν το, το σε στόχο, να κερδίσει τις εκλογές. Ποιος στέει, το ευρωπαϊκό σύστημα που επιτρέπει την διαφθορά δίνοντας επιδοτήσεις στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αντί να αφήσουμε την αγορά και τους κανόνες της αγοράς, έχουμε ένα σύστημα εξάρτησης από τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διονύζεται. Και το να αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά πολιτικά είναι ε, ίδιον των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Αμαρζή, πρόεδρε. Επίτροπε, ας το πούμε απερίφραστα. Υπάρχει διαφθορά για τα ευρωπαϊκά κονδύλια και μία. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης θέλω να σας πω ότι ένας αγώνας αμήλικτος πρέπει να γίνει κατά της διαφθοράς ε, εναντίον των διαφθορτικών ταμείων. Είναι θέμα αξιοπιστίας των πολιτικών μας και είναι θέμα εμπιστοσύνης στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σε αυτόν τον αγώνα θα μας βρείτε, θα με βρείτε στο πλευρό σας, όπως θα με βρείτε και θα μας βρείτε στο πλευρό σας, ούτω ώστε να δοθεί συνέχεια στη σύγκρουση συμφερόντων και στο τεκμήριο ε, απάτης, αν όχι διαφθοράς, στην τσεχική δημοκρατία. Έχουμε τώρα μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γιατί τη φτιάξαμε για να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ε, η επικεφαλής της αγγελίας διορίστηκε και τι μαθαίνουμε, ότι δεν έχει τα απαραίτητα μέσα για να διεξάγει αυτόν τον αγώνα που πρέπει να διεξαχθεί όμως. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να προσπαθήσουμε για να υπάρχει δημοσιονομική ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι πραγματικά ανεξάρτητη και θα υλοποιήσει τους στόχους της μόνο αν έχει τα μέσα, οικονομικά μέσα δηλαδή, για να μπορέσει να κάνει αυτό το βασικό αγώνα κατά της διαφθοράς. Διαφθοράς ε, εναντίον των διαφορετικών ταμείων και της ΚΑΠ για να προστατεύσουμε τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Η πρόεδρος ε, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, κυρία Χόλμαγερ, έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, ε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, συνάδελφοι, για πρώτη φορά η συζήτηση αυτή, κυρία Καράντσοβα, δεν είναι εσωτερική τσεχική συζήτηση. Ε, έχει να κάνει αυτό και με την παρέμβαση της κυρίας παντέλε Δεν ε, μας ενδιαφέρει τι γίνεται εντός της ε, Τσεχίας. Ε, δεν αφιζητούμε καμία δικαστική διαδικασία. Αλλά έχω δύο ερωτήσεις και παρακαλώ η Κομισιόν και το Συμβούλιο να με στηρίξουν. Πρώτον, η ευρωπαϊκές ενισχύσεις δεν επιτρέπεται να στηρίζουν ολιγαρχικές δομές. Ε, υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ε, και υπάρχει το άρθρο 81. Πρόκειται για νομοθεσία κατά των ε, ολιγαρχών. Και το δεύτερο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι πόσε ευρωπαϊκέ ενισχύσει επιτρέπεται ένα πρόσωπο να λάβει εντό ενό έτου και ενό εντός δημοσιονομικού πλαισίου. Διότι χάνουμε την αξιοπιστία μα εάν ένα πρόσωπο λαμβάνει 100, 200, 300 εκατομμύρια και κάποιο άλλο λαμβάνει μόλι 5.000. Ε, δεν ε, είναι δίκαιο αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ιντσίρ ε, κύριε Πρόεδρε, ε, η επανάληψη της ε, ποινική διαδικασίας κατά του Πρωθυπουργού της Τσεχίας είναι σημαντική. Δεν επιτρέπεται τα χρήματα των φορολογούμενων πολιτών να χρησιμοποιούνται για απάτες. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και γι' αυτό είναι σημαντικό να συζητάμε την διαφθορά που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Δυστυχώ, ο Πρωθυπουργός της Τσεχίας ε, είναι μόνο ένα παράδειγμα. Η διαφθορά, η απάτη, η κατάχρηση κονδυλίων ε, είναι φαινόμενα σε πολλά μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωση. και γνωρίζουμε ότι είναι κάτι που εμποδίζει την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και γι' αυτό είναι υψής της σημασίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει στα σοβαρά υπόψη την, ε, το καθήκον της ε, ως ελεγκτή. Η Ευρώπη θα πρέπει να βασίζεται στη δικαιοσύνη ε, και την κοινωνία. Οι κοινοί μας πόροι δεν επιτρέπεται να καταλήγουν στις τσέπες διαφερμένων προσώπων. Μηδενική ανοχή και μόνο έτσι θα καταφέρουμε να κρατήσουμε ενωμένη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κνότεκ. Ευχαριστώ. Ο Πρωθυπουργό Μπάμπη ξεκίνησε το 2011 ε, με την πλατφόρμα του κατά της διαφθοράς. Οι ενισχύσεις που δόθηκαν ε, ήταν ε, κάποια από τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι πραγματικές διαδικασίες ξεκίνησαν ε, το 2015. Ε, πέρυσι όμως ε, σταμάτησαν διαδικασίες δίωξής του, μετά δόθηκαν και άλλες πληροφορίες και συμμετείχε η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη. Είναι σαφής η πολιτικοποίηση του θέματος αυτού. Ε, τελικά οι εταιρείε του Πρωθυπουργού μπήκαν σε ένα καταπίστευμα. Πρέπει να δούμε ε, πώς ορίζεται αυτή η σύγκρουση συμφερόντων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει, νομίζω, μια επιβλαβή πολιτική συζήτηση. Κύριο Πέξα. Πρόεδρε, συνάδελφοι, σε μια συζήτηση για την Πολωνία και την ε, Ουγγαρία. Τι να πει κανεί και εδώ καινούριο. Ο κύριος Μπάμπης δεν είναι η μόνη περίπτωση. Ε, η όλη κατάσταση και οι μηχανισμοί ελέγχου των οικονομικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. Ο κύριος Μπάμπης απλώς κατάφερε να δημιουργήσει ένα καταπίστευμα με τι εταιρείες του και να παρακάμψει τον όλο μηχανισμό. Είναι λοιπόν ε, ένα γνωστό τρίκ που χρησιμοποιούν κάποιοι από τους κυβερνώντες ε, και κάνουν αυτό που θέλουν. Αλλά δούμε και το άλλο σκέλος. Είναι ιδιοκτήτης μιας από τις μεγαλύτερες, ενός από τους μεγαλύτερου οικονομικού ομίλου στην Δημοκρατία της Τσεχίας και παίρνει ένα τεράστιο μερίδιο ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το χρησιμοποιεί για να αυξήσει την επιρροή του εντό τη χώρα και να διατηρήσει τη θέση του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της εταιρεία του, τη Αγκροφέρτ, ε, χρηματοδοτεί απευθεία τη δική του πολιτική εκστρατεία εκ μέρους ε, των βουλευτών του και άλλων αυτών δεν προστατεύει μόνο τον ίδιο, ούτε εξυπηρετεί μόνο τον ίδιο, αλλά και όσου έχουν διαπλεκόμενα συμφέροντα μαζί του ε, ή και σε άλλε χώρε. Οπότε, όταν μιλάμε για σοβαρά μέτρα, πρέπει να υπάρξει βεβαίω ομοφωνία. Όμω αυτοί οι ολιγάρχε υπερασπίζουν ένα τον άλλο, οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εναντίον του. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Μπλάσκο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, συνάδελφοι, οι πολίτες της Δημοκρατίας της Τσεχίας έχουν μπουχτίσει με τις αλλεπάλληλες συζητήσεις για τα προβλήματα που προκαλεί ο κύριος Μπάμπης. Και όσο πιο πολύ συζητάμε για τα ζητήματα αυτά, τόσο πιο πολύ τον υποστηρίζουν και άλλοι ψηφοφόροι. Ας αφήσουμε το θέμα στους ε, Τσέχους, τους ίδιους να το αποφασίσουν ε, και στις τσεχικές αρχές. Δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να ε, πει ξεκάθαρα και με βεβαιότητα στον κύριο Μπάμπη, είστε ένοχο για κάτι. Είναι εσωτερικό ζήτημα τη Τσεχία και του δικαστικού τη συστήματο, των δικαστηρίων. Έχουμε άλλα σοβαρότερα ζητήματα να συζητήσουμε εδώ πέρα. Όχι αυτό. Το κοινοβούλιο μα είναι υπέρ τη ισότητα των φίλων. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω να συσταθεί επιτροπή που θα ερευνήσει τις δραστηριότητες, τις Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φοντερ Λάιεν. Διότι και εκείνη είναι υποπτή για ε, υποθέσεις σύγκρουση συμφερόντων στη δική της τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να κάνει την απαραίτητη έρευνα ε, και να υπάρξει και απάντηση για τις πολιτικές ευθύνες του καθενός. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Φλάναγκαν. Ευχαριστώ. Υπόθηκε προηγουμένως από κάποιον εδώ ε, ότι Υπάρχει εδώ θέμα προκατάληψη. Από τη δική μου πλευρά δεν υπάρχει καμία προκατάληψη. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι εάν υπάρχει υπεξαίρεση, θέλουμε πίσω τα λεφτά. Ο κόσμο έχει βγει στου δρόμου και ε, έχει διαδηλώσει. Δεν έχουν αρκετά για να πληρώσουν του φόρου του. Και εμεί εδώ έχουμε εκλεγεί για να, βοηθ... βεβαιωθούμε ότι το χρήμα πηγαίνει σε αυτού που πρέπει. Ε, το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο με την υποστήριξη τη Γεωργία και τα διευθυντικά ταμεία έχει δώσει πολλέ δυνατότητε. Αλλά δυστυχώ έχουν χάσει την εμπιστοσύνη του Ευρωπαίοι πολίτε, διότι δεν βλέπουν να πηγαίνουν τα χρήματα στου στους πραγματικού δικαιούχου. Ε, έτσι δεν έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και δεν μπορούμε να επαφιόμαστε μόνο στα κράτη-έθνη όπω παλιά. Πρέπει όμω να δημιουργήσουμε το κατάλληλα αρχιτεκτόνημα ώστε μέσα από το σωστό διάβλο τα, τα χρήματα να πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Διότι αυτή τη στιγμή τα χάνουμε και δεν ξέρουμε πού πηγαίνει τι είτε παρανόμω είτε νομίμω, θα πρέπει να ξέρουμε πού έχει πάει το κάθε τι και να μπορούμε και να τα ανακτήσουμε όταν πρέπει. Ευχαριστούμε, κύριο Μουρισάνη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, ε, κύριε Υπουργέ. Ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχεται από χρήματα που πληρώνουν οι πολίτε και γι' αυτό είναι καθήκον μα ω μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υπερασπιστούμε του πόρου αυτού και να του δαπανίσουμε ε, με καλό τρόπο. Οποιαδήποτε κατάχρηση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαράδεκτη, πόσο μάλλον όταν γίνεται από Πρωθυπουργό. Ε, είναι απαράδεκτο αυτό και τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, πρέπει να ανακτήσουμε τους πόρους ε, και να φροντίσουμε να επιστραφούν όλα τα ποσά αυτά στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό έχουμε τον Όλαφ και γι' αυτό δημιουργήσαμε ε, και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να είναι ισχυρή και ανεξάρτητη και να μπορεί να ενεργεί σε τέτοιε περιπτώσει. Ε, σημαντικό είναι η κυβέρνηση του κυρίου Μπάμπη να επιστρέψει τα ε, ποσά αυτά και όχι οι πολίτε να πρέπει να πληρώσουν. Και αν υπάρχει ποινικό αδίκημα, θα πρέπει να γίνει σωστή έρευνα. Και πέρα από, δικαστικ... πέρα από τι δικαστικέ συνέπειε, Υπάρχει και πολιτική ευθύνη ε, του κόμματος ε, ε, του κυρίου Μπάμπης καθώς και του, της πολιτικής του ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του Ρινιού. Ευχαριστώ συνάδελφε, ο κύριος Λιμπεράτσκι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπε, έχω την εντύπωση ότι το Συμβούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι δική του υπόθεση. Ο Επίτροπος παρουσίασε όλη τη διαδικασία και προς το τέλος της ομιλίας του ανέφερε ότι η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 24 ακόμη μήνες. Αυτό όμως το χρονικό διάστημα είναι υπερβολικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι κάνει. Ζητάει δράση. Περί χρημάτων πρόκειται δεν είναι πολιτικό θέμα. Τα χρήματα δαπανούνται σωστά ή υπάρχει κατάχρηση κοντιλίων. Αν υπάρχει κατάχρηση κοντιλίων θα πρέπει να επιστραφούν. Και αυτό δεν είναι απόκειται στα τσεχικά δικαστήρια να το αποφασίσουν αυτό, αλλά τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να λάβουν σχετική απόφαση. Ε, μας λέτε τώρα ότι είναι ικανός επιχειρηματίας ο κύριος Μπάμπης. Ε, τρέχα γύρευε δηλαδή. Ο κύριος Ιώχημ Κούς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευγνώμων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ε, ε, έχει παρουσιάσει θέση σχετικά επιφρακτική όσον αφορά την υπόθεση αυτή του κυρίου Μπάμπης ε, τη στιγμή που ακόμη διεξάγονται οι έρευνες. Οι έρευνες αυτές θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν προτού καταδικάσουμε κανέναν. Εάν δεν το κάνουμε αυτό τότε αυτομάτως ε, θα μας κατηγορήσουν ε, ότι ε, η συζήτησή μας βασίζεται σε ζήλια. Δεν... Θέλουμε ο κύριος Σεμπάμπης να έχει επιχειρήματα σε υποθέσεις όπως είναι η μετανάστευση, η διατήρηση του σεχικού νομίσματος κλπ. Θα πρέπει να είμαστε ουδέτεροι και να περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και να αναρωτηθούμε εάν οι κανόνες μας είναι κατάλληλοι ή εάν θα πρέπει να καταργήσουμε τελείως τις ε, επιδοτήσεις. Ευχαριστώ, Σαρβάμα. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ακούσετε όλοι σας πολύ προσεκτικά και εσείς Κομισιόν. Είναι πολύ επιβλαβές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό εδώ είναι καταστροφικό για τη δημόσια εικόνα της Ένωσης. Θεωρητικά, η περίπτωση Μπάμπης δεν είναι καν η μοναδική περίπτωση τέτοιου τύπου. Ξέρουμε όλοι τι συνέβη σε άλλη χώρα. Δεν θέλω να μιλήσω καν για τον Μπάμπης. Θέλω να πω το εξής. Αν οι δημοσιονομικοί κανονισμοί και το άρθρο 61 δεν είναι επαρκέ, θα πρέπει να το αλλάξουμε. Και θα πρέπει να το αλλάξουμε το δημοσιονομικό κανονισμό γρήγορα, αν δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε πραγματική εξουσία εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να έχει του απαραίτητου πόρου για να κάνει το έργο τη. Ευχαριστούμε. Προ στιγμήν δεν βλέπω τον επόμενο αγορητή στην αίθουσα τον κύριο Τσουχονταρού. Οπότε, εάν δεν εμφανιστεί, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βίντσικ, που είναι επικεφαλής αντιπροσωπής του ΕΛΚ. Την κυρία Βίντσικ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η απάτη και η διαφορά δεν έχουν θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τους φορολογουμένους της Ένωσης. Εδώ βλέπουμε ότι ο κύριος Ντάβιντ βέβαια έχει φύγει από την αίθουσα. Βλέπουμε κάποιοι να λένε ότι το θέμα είναι εσωτερικό της χώρας. Εδώ όμως αυτό δεν είναι απλώς εσωτερικό, είναι θέμα μιας επιχείρησης που έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Εγώ θα ζητούσω δημοσίως να αναλάβουν τα θεσμικά όργανα το ρόλο τους και να μην υπάρχουν τέτοιου είδους παραγραφές. Για ένα πολιτικό οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι ε, όχι απλώς ε, οικονομικές αλλά και ηθικές. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε δύο μέτρα και δύο σταθμά εντός της ίδιας ομάδας. Θα πρέπει λοιπόν να διαλευκανθεί η υπόθεση και να δούμε αν μπορεί να επιστραφούν τα ποσά, αυτά. Θα πρέπει οι πολιτικές συνέπειες να μην ε, βαρύνουν άλλο τους πολίτες της χώρας και να δημιουργούν προβλήματα για το μέλλον τους. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόβλημα εδώ δεν είναι μόνο ένα μεμονωμένο κράτος μέλος. Το έχουν γράψει αυτό και οι New York Times η περιφερειακή ανάπτυξη και τα διευθυντικά ταμεία δεν είναι ε, κονδύλια που πρέπει να πηγαίνουν στο πορτοφόλι των ολιγαρχών, αλλά στις οικογένειες των φορολογουμένων. Θέλουμε λοιπόν να δούμε πολύ σοβαρά την πρόταση του Επιτρόπου Χόγκαν, την υποστηρίζω, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα κάπινγκ, ανώτατα όρια δηλαδή, και να εφαρμόζονται αυτά, διότι τα ποσά αυτά θα πρέπει να υποστηρίζουν οικογενειακές επιχειρήσεις, όχι οικογένειες της ελίτ ή κάποιων ολιγαρχών. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε να μην βασιζόμαστε απλώς στην καλή προαίρεση και σε όσα λέγονται, αλλά να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και όταν υπάρχουν παραβιάσεις θα πρέπει να βαρώνται και κατάλληλε τιμωρίε. Κυρίε και κύριοι, θεωρώ λογικό να καθυστερήσει η υπόθεση Μπάμπης. Ο Μπάμπη είναι ο μεγαλύτερο ε, δικαιούχο ε, χρημάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προ την Τσεχική Δημοκρατία. Είναι λεφτά των φορολογουμένων. Επομένω είναι απόλυτα λογικό οι ευρωβουλευτέ και οι εκπρόσωποι να θέλουν τη Ευρώπη να κάνουν μια συζήτηση για αυτό το θέμα. Δεν είναι λογικό, φυσιολογικό, ένα από του πλουσιότερους τσέχου να παίρνει λεφτά τα οποία προ... προορίζονται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για φτωχές περιφέρειες. Ας εξασφαλίσουμε ότι θα διερευνηθεί σωστά η υπόθεση αυτή. Οι Τσέχοι πολίτες θέλουν να γνωρίζουν πολύ ακριβώς τι υπάρχουν σε αυτές τις ε, ελεκτικές εκθέσεις. Τι κάνει ο Πρωθυπουργό, αν παραβιάζει τον νόμο και πόσο μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει γύρω του. Τώρα, αν είναι υπεύθυνο, θα αποφασίσει η τσεχική δικαιοσύνη. Αλλά σε εξασφαλίσουμε ότι ποτέ πια οι ολιγάσεις δεν θα παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Και τώρα ξεκινάμε το Catch the Eye. Έχω ένα αίτημα από την κυρία Σόιντροβα. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο, συνάδελφοι. Είμαι από την Τσεχία και ως Ευρωβουλευτής από την Τσεχία, από την Τσεχία δεν θέλω να συζητάμε και στην υπόθεση Μπάμπη. Απ' την άλλη καταλαβαίνω και τους συναδέλφου, οι οποίοι θέλουν να υπάρχει έλεγχο των Ευρωπαϊκών ε, Ταμείων. Μετά από έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων γύρω από το πρόσωπο του Πρωθυπουργού της Τσεχίας και ότι υπάρχει κατάχρηση κονδυλίων τη Ευρώπη. Τα λεφτά που δόθηκαν στο project αυτό Storks Nest, την φωλιά του πελαργού, ε, επιστράφηκαν στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και επομένω δεν υπάρχει ω προ αυτό ζημία ε, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό ούτε στον εθνικό προπολογισμό. Αλλά εγώ θυμάμαι τα πρώτα λόγια του κύριου Μπάμπη, ο οποίο είπε το εξή. Παραθέτω. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το project αυτό, με τη φωλιά του πελαργού. Δεν έχω ιδέα γι' αυτό. Και μόνο μετά τι έρευνε θυμήθηκε ξαφνικά. Έφνης ο κύριος, ότι του ανήκε. Εμείς δεν κρίνουμε. Θέλουμε απλώς μία ενδελεχή έρευνα γιατί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να προστατεύεται και δεν πρέπει να υπάρχουν καταχρήσεις βάρος του. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφε. Ο Επίτροπος Συρκεβίσιους έχει το λόγο. Let me conclude, first of all, by stressing... Ευχαριστώ να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μηδενική ενοχή για την απάτη, την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ξέρω ότι το σώμα αυτό υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην καταπολέμηση τη απάτη και σε ό,τι αφορά τα διαφορετικά κονδύλια. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το δημόσιο χρήμα δαπανάται όπω δει να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση τον Μάιο του 2018 για την προστασία του ευρωπαϊκού προπολογισμού σε περίπτωση γενικών ατασταλιών ή παρατυπιών σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου στα κάτι μέλη. Η πρόταση προβλέπει μηχανισμό για την, ε, ανα... για την αναστολή ή την ανάκτηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση του κάτω δικαίου. Το... Αυτό συνέβη στην εφαρμογή του ελεγκτικού μηχανισμού για τις καταγγελίες ε, επεξαιρέσεις ε, κονδυλίων, το δικαστικό σύστημα, η αυθαίρετη επιβολή νόμου, οι αυθαίρετες αποφάσεις των δημόσιων αρχών μπορεί να ε, περιορίσουν την σωστή άσκηση ένδικων μέσων τέτοιοι περιορισμοί για την πραγματική έρευνα, διαλεύκανση, εξερεύνηση, διερεύνηση μάλλον και επιβολή ποινικών ευθυνών είναι τέτοιες περιπτώσεις. Πρέπει να σεβόμαστε τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Έχουμε μηδενική ενόχη για την κατάχρηση κονδυλίων και έχουμε καταγράψει τι κατηγορίε για υπεξαίρεση χρηματικών ποσών στην Δημοκρατία τη Τσεχία. Πρέπει να προστατεύσουμε τον προπολογισμό και έχουμε λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Δεν μπορεί να ε, χρηματοδοτούνται έργα που έχουν σχέση με την υπόθεση της ε, σύγκρουση συμφερόντων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει τα ποσά που μπορεί ε, να ε, αφορούν την υπόθεση αυτής τη σύγκρουση συμφερόντων και ε, για το αν θα ανοίξει και πάλι όχι η ποινική διαδικασία κατά του κ. Μπάμπη, η εθνική ε, δικαστική διαδικασία είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των τσεχικών αρχών. Οι τσεχικέ αρχέ ερεύνησαν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει καμία ε, συνέπεια για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σα στηρεί ενήμερου. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε. Και τώρα, εξ ονόματος της, ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Υπουργός Μπρνιάτς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Να θυμίσω πόσο σημαντικό είναι για το Συμβούλιο ε, να προστατεύεται οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και να διαπιστώνει ότι το δημόσιο χρήμα δαπανάται ε, με νόμιμους τρόπους. Είναι βέβαια ευθύνη του Εθνικού, ευθύνη του Εθνικού Εισαγγελέα και των δικαστών το να ελέγξουν την υπόθεση εσωτερικά και βεβαίω σύντομα θα είναι θέμα και τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καταγράφω τι ανησυχίε σα καθώ και του δείκτε που μα ανέφερε ο Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την ε, Υπουργό. Κλείνει η συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα γίνει στην Σύνοδο του Φεβρουαρίου. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την 15η Σύνοδο τη Διάκριση των Μερών, COP15, τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα. Θυμίζω, συνάδελφοι, ότι μπορείτε και να εγγραφείτε ω συνήθω, είτε με ηλεκτρονικά μέσα για την διαδικασία ΚΑΤΣΔΙΑ και για τι γαλάζιε κάρτε. Τι οδηγίε θα τι βρείτε σε έντυπο που βρίσκεται στην είσοδο τη Ολομέλεια. Τώρα να δώσω το λόγο του ονόματο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Επίτροπο Σινκεβίτσιου. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, το Νοέμβριο το Κοινοβούλιο ε, ε διακήρυξε ε, το θέμα του κλίματος ε, ως επίγον. είδαμε ξηρασία, είδαμε ακραία καιρικά φαινόμενα, είδαμε τεράστια μείωση των επικονιαστών και όλο αυτό δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για άμεση δράση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε σοβαρά υπόψη το θέμα αυτό και μια από τις πρώτες αποφάσεις ήταν ε, η Πράσινη Συμφωνία, νέα, ε, νέο θεματολόγιο για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστούν ε, οι πιο σημαντικές προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγείται όσον αφορά την ουδετερότητα ως προς το κλίμα και στόχος είναι στο Κουνμίν το 2020 να συμφωνήσουμε πάνω σε ένα πλαίσιο για τη βιολογική ποικιλότητα. Επικροτώ το ότι το Κοινοβούλιο στηρίζει απόλυτα τη φιλοδοξία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ηγηθεί, ε, να αποτελέσει υπόδειγμα. Η στρατηγική βιοπικιλότητα 2030 ε, που θα υιοθετήσουμε μέχρι τον Μάρτιο του 2020 θα συμπεριλαμβάνει ε, προτάσεις για δεσμευτικά μέτρα και στόχους. Οι προετοιμασίες ε, γίνονται αυτή τη στιγμή εντό Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ψήφισμα που υιοθετήσετε εσεί αύριο θα αποτελέσει σημαντική έμπνευση και για τους προβληματισμούς ε, μας και για τις φιλοδοξίες μας. Ε, δεν επιτρέπεται να ξανααποτύχουμε όσον αφορά τους στόχους βιοπικιλότητας. Οι επιστήμονε είναι απόλυτα σαφή, χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε ε, την περιβαλλοντική και ε, κλιματική επίγουσα κατάσταση. Ε, μετά το 2020 όσον αφορά το πλαίσιο βιοπικιλότητας. Στηρίζουμε το Ευρωκοινοβούλιο ε, στο αίτημά του για έναν πιο αποτελεσματικό μηχανισμό. Χρειαζόμαστε έναν συστημικό και τακτικό κύκλο για αναθεώρηση της ε, προόδου ε, για να μειωθούν οι πιέσεις όσον αφορά την βιοπικιλότητα. Ε, χρειαζόμαστε έναν στόχο ανάλογο με αυτόν του 1,5 βαθμού Κελσίου για το κλίμα. Και θα πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα τον κύκλο αυτών ε, θα πρέπει μέχρι το 2021 να μπορούμε να ελέγξουμε τις δράσεις, ώστε το 2022 να μπορούμε να αναθεωρήσουμε τις δράσεις μας στους πιο σημαντικούς τομείς. Τέλος, το πλαίσιο δικτών και παρακολούθησης θα πρέπει να περιλαμβάνει δείκτες που να μας επιτρέπει αξιολόγηση των εθνικών συνεισφορών για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων θα ήθελα να τονίσω τις συνέργειες ε, με την διακυβέρνηση των ωκεανών και τις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται για νέα, δημοσ... για νέα διεθνή σύμβαση για τον νόμο των θαλασσών. Είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε τα μέσα για την υλοποίηση ε, των στόχων αυτών. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διπλασιάσει την ε, χρηματοδότηση για τη βιοπικιλότητα προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Θα πρέπει να κινητοποιήσουμε εσωτερικούς πόρους και θα ήθελα να τονίσω τρεις σημαντικές πτυχές εδώ πέρα. Πρώτον, ο κόσμος συνεχίζει να δαπανεί περισσότερα χρήματα για τη διόρθωση ε, της βιοπικιλότητας από ό,τι σε προορατική δράση. Χρειάζεται να αναμορφώσουμε τις ε, πολιτικές μας ε, ώστε να διασφαλίζεται η βιοπικιλότητα. Δεύτερον, η αποκατάσταση οικοσυστημάτων είναι πιο ακριβή από τη διατήρηση. Όσο πιο γρήγορα προστατεύσουμε την φύση και αποφύγουμε την απώλεια βιοπικιλότητα σε τόσο ε, λιγότερες διορθωτικές δράσεις θα χρειαστούν. Και τρίτον, ε, θα πρέπει να αυξήσουμε τις ε, επενδύσεις σε λύσεις για τον μετριασμό του, της αλλαγής του κλίματος, την, διατροφική, την επιστημιστική ασφάλεια και την υγεία. Χρειάζονται ισχυρές δεσμεύσεις για να προστατεύσουμε καλύτερα τις ε, περιοχές πλούσιες σε βιοπικιλότητα για να αποκαταστήσουμε ε, οικοσυστήματα και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ε, με βιώσιμο τρόπο τους πόρους μας. Και θα πρέπει ε, η βιοπικιλότητα να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές μας ε, και στις πιο απόμακρες περιοχές. Θα πρέπει να φροντίσουμε να ε, τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας δημιουργώντας ένα πλαίσιο που να μας επιτρέπει επίτευξη των στόχων μας. Πρέπει να αποκαταστήσουμε την φύση, την βιοπικιλότητα και παρέχοντας επαρκή χρηματοδότηση. Το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα είναι ζωτική σημασία. Ε, θα πρέπει να διασφαλιστούν επαρκεί πόροι για την προστασία, ε, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση οικοσυστημάτων. Ε, έχουμε την κοινή γεωργική πολιτική, την πολιτική συνοχή και τα διαρθρωτικά ταμεία. Ορίζον έχουμε τα προγράμματα ορίζων και άλλα και θα πρέπει να φροντίσουμε η χρηματοδότηση αυτή να αποτελέσει μοχλό και για η ιδιωτική χρηματοδότηση. Θα πρέπει να φροντίσουμε οι αλλαγέ αυτές να μην αφήσουν κανέναν πίσω. Θα πρέπει να στηρίξουμε τους ε, γεωργούς μας, ε, τους ε, δασοκόμους, τους αλληλεί κατά τη μετάβαση αυτή. Επίσης θα πρέπει να αποφύγουμε Ε, να καταναλώνουμε προϊόντα τα οποία δεν παράγονται με βιώσιμο τρόπο. Γι' αυτό η στρατηγική μας θα πρέπει να ασχοληθεί και με την βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή. Ε, θα πρέπει να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα και η βιοπικιλότητα να ε, ληφθεί υπόψη και στην εμπορική πολιτική μας. Θα πρέπει επίσης να έχουμε καλύτερη συνεργασία με του διεθνεί μα εταίρους θα πρέπει ε, να υπάρχουν εργαλεία ώστε να λογοδοτούν ε, οι άλλες χώρες όσον αφορά την βιοπικιλότητα τους. Ε, το παράθυρο ευκαιρίας για να πετύχουμε τους στόχους μας όσον αφορά τη βιοπικιλότητα, για να ζούμε σε αρμονία με τη φύση, κλείνει γρήγορα και τα επόμενα χρόνια θα είναι κρίσιμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά ε, τι ευθύνη έχει κατά διάρκεια αυτή τη πενταετού θητεία. Ε, μπορείτε να βασιστείτε στην προσήλωσή μα για να πετύχουμε του κοινού μα στόχου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άτσου Λαμπαγέ, στη γλώσσα του Επιτρόπου. Και τώρα ξεκινούμε με τις παρεμβάσεις από τις πολιτικές ομάδες. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η κυρία Ευγόν, 1,5 λεπτό. Αγαπητή Ανιές, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο ΙΕ τη Δευτέρα πρότεινε να προστεύσουμε το 30% του πλανήτη μέχρι το 2030. Η COP15 προωθεί 17 στόχοι, στόχους για να ε, περιορίσουμε την επίπτωσή μας στην φύση, για να συνδέσουμε το κλίμα με τη βιοποικιλότητα που είναι οι δύο όψεις ενός νομίσματος και έχουν να κάνουν την επιβίωση του πλανήτη. Συμφωνώ απολύτως με τους στόχους αυτούς. Αντίθετα από παλιά ευχολόγια, ε, τώρα έχουμε συγκεκριμένους ε, στόχους με αριθμούς, με τρόπους για να τους υλοποιήσουμε. Με αυτό, αυτό ακριβώς υποστηρίζουμε και στο ψήφισμά μα. Αλλά και πάμε και πιο μακριά. Θέλουμε αυτή η στόχη να είναι νομικά δεσμευτική, ούτω ώστε να μην μείνουν γράμμα κενό περιεχομένου. Η COP15 θα πρέπει να είναι κάτι το αντίστοιχο με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Από τώρα θα πρέπει να δράσουμε πολύ συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη στρατηγική που θα παρουσιάσει το Μάρτιο να λάβει ήδη και να προωθήσει τέτοιου ε, υποχρεωτικού στόχου και να ε, εντείνει του στόχου όλε τι πολιτικέ. έχουμε περισσότερη έρευνα και κοινοτομία. στηρίξουμε μαζικά τους αλείς και τους γεωργού, καθώς και τους δασοκόμους για να έχουν πρακτικές πιο βιώσιμες. Οι υπεύθυνοι είναι και τα κράτη-μέλη, αλλά και κάθε δήμος και κοινότητα. Ας μην περιμένουμε τον Οκτώβριο. Τώρα πρέπει να δράσουμε. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, συνάδελφε. Και τώρα, από τους σοσιαλιστές... Για μισή λεφτά ο κύριος Λουένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την παρουσίασή του. Καταρχάς, θα ήθελα τώρα που μιλάμε για την καταπολέμηση της αλλαγής του πλανήτη για την προστασία της ε, βιοπικιλότητας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ε, επιστήμονες, γιατί αυτοί αφυπνίζουν τον κόσμο και γιατί υπάρχει μια δέσμευση από την επιστήμη και τους οικολόγους. Από το 1900 μειώθηκε το προσδόκιμο ζωής κατά 20% για όλους τους ζώντες οργανισμούς. Ε, για τα αμφίβια, περίπου το 33% από, τα, ε, από τους κορολαγενείς φράχους και το 1 τρίτο όλων των θαλάσσιων θηλαστικών απειλούνται είναι η έκτη μαζική ε, καταστροφή ζώων των οργανισμών. Τι άποψη έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 96% των ε, επιστημόνων λένε ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τη φύση. Και ποιος έχει την ευθύνη. Όλοι μας. Να προστατεύσουμε τη ζωή και τον πλανήτη και να ζητήσουμε να, ακούσουμε τους πολίτες. Αυτό είναι η προτεραιότητα των σοσιαλδημοκρατών. Και αυτό προτάσουμε σε αυτό το ψήφισμα. Έφτασε μία πολύ γρήγορα. Η οικολογική μετάβαση θα πρέπει να είναι δίκαιοι, αγαπητοί φίλοι. Δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν νέε ανισότητε. Ε, φορολογική, περιβαλλοντική μάλλον φορολογία. Χρειαζόμαστε επαρκεί πόρου. Ένα φορολογικό μοντέλο σωστό. Όποιο ε, ρηπαίνει περισσότερο θα πρέπει να πληρώνει περισσότερο. Η αποψήλωση των δασών. Θα πρέπει να έχουμε νομοθεσία ούτω ώστε να καταπολεμήσουμε την αποψήλωση. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει παράνομη υλοτόμηση των δασών. Αυτά θα πρέπει να είναι δεσμευτικά όμω, αγαπητό ΑΕΛΚ. Αλλιώ δεν θα πετύχουμε τίποτα. Είναι σημαντικό επίση να αυξήσουμε τι ε, προστατευόμενε ε, ζώνε. 30% τώρα και μέχρι το 2050 50%. Και να μειώσουμε το ποσοστό των ε, φυτοφαρμάκων. Να συμφωνήσουμε για ένα ποσοστό μείωση των φυτοφαρμάκων. Δεν έχουμε άλλο πλανήτη. Ένα είναι. Ένα ανήκει στου ανθρώπου. Εδώ ζούμε. Εδώ βρισκόμαστε. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό απέναντι στα έμβια όντα του πλανήτη αυτού και στην βιοπικιλότητα να τον προστατεύσουμε. Ε, θα πρέπει λοιπόν να πάμε στην Κίνα με μία ενιαία φωνή και να προστατεύσουμε την βιοπικιλότητα και τον πλανήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Grazie σε διάφορες γλώσσες. Και τώρα, Ροντρίγκες Ράμος από το Renew Europe. Για δύο λεφτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει προκλήσεις περιβαλλοντικές σαν προηγουμένου. Η απώλεια βιοπικιλότητας είναι μία από τις προκλήσεις. Όπως υπόθηκε ήδη, γινόμαστε μάρτυρες μιας κατάστασης που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επίγουσα ανάγκη, γιατί το 70% των χερσαίων οικοσυστημάτων και το 40% των θαλάσσιων οικοσυστημάτων βρίσκονται σε μία κατάσταση επιδείνωσης και κινδύνου. Μπαίνουμε σε μία φάση που θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε η έκτη μαζική καταστροφή ζών των οργανισμών και η καταστροφή του περιβάλλοντος. Γιατί ο αριθμός των ειδών που εξαλείφονται είναι μεγαλύτερος από ό,τι εξαλείφθηκε σε όλη την υπόλοιπη ανθρώπινη ιστορία. Θα πρέπει να δράσουμε λοιπόν ενώπιον αυτών των προκλήσεων. Και αυτό κάνουμε με αυτό το ψήφισμα ως Κοινοβούλιο. Ζητάμε από την Κομισιόν μεγαλύτερη φιλοδοξία και μια νέα στρατηγική για την προστασία της βιοπικιλότητας. Και αυτή η μεγαλύτερη φιλοδοξία και αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική θα πρέπει να είναι το επισκεπτήριό μας στην επόμενη συνεδρίαση της COP15 στην Κίνα. Θα πρέπει να έχουμε δεσμευτικούς στόχου για να προστατεύσουμε, προστατεύσουμε τις ε, φυσικές περιοχές 30% μέχρι το 2030 και το 50% το 2050, το μισό του πλανήτη. Δεσμευτικούς στόχους για να αποκαταστήσουμε ζώνες που έχουν ε, επιδεινωθεί πάρα πολύ και οικοσυστήματα που κινδυνεύουν από εξαφάνιση. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε περισσότερα χρήματα. Δεν μπορούμε να έχουμε περισσότερε φιλοδοξίε με λιγότερα χρήματα. Ένα 10% του νέου πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να δοθεί ειδικά για την προστασία τη βιοπικιλότητα. Και επίση θα πρέπει να δουλέψουμε μαζί με όλους τους φορείς που έχουν να κάνουν και συνδέονται με αποφάσει για την προστασία τη βιοπικιλότητα. Γεωργούς, και αλής. Αυτή είναι εταίρη μας. Κανένα στόχος τη συμφωνίας του Παρισιού, της ε, πράσινη συμφωνία δεν θα το πετύχουμε εάν δεν είμαστε φιλόδοξοι σε αυτή τη νέα στρατηγική για τη βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Και τώρα εκ μέρους των ε, Πρασίνων ο κύριος Νίνιστερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η βιοπικιλότητα παγκοσμίω απειλείται. Δεν καταστρέφουμε απλώς ε, τις συνθήκες διαβίωσης για μας με τις κλιματικές αλλαγές που προκαλούμε, αλλά κατασπαταλώνται και οι φυσικοί πόροι. Ο τρόπος που παράγουμε τα τρόφιμά μας επηρεάζει συνολικά το μέλλον του πλανήτη και της βιοπικιλότητάς του. Την χλωρίδα και την πανίδα. Κορυφαίοι επιστήμονε μα είπαν ότι ένα εκατομμύριο ήδη ω το 2030 θα έχουν εξαφανιστεί από τον πλανήτη αν δεν αλλάξουμε την συμπεριφορά μα. Είναι σαφέ λοιπόν ότι η Σύνοδο για τη ποικιλότητα πρέπει να γίνει ένα ε, γεγονό ανάλογο με τη Σύνοδο του Παρισιού για το κλίμα. Πρέπει να βρούμε δεσμευτικού στόχου, διότι όσοι έχουμε κάνει ω τώρα παγκοσμίω δεν έχουν επιτευχθεί. Ε, πρέπει να υπάρξει μια νομικώ δεσμευτική διαδικασία που να επιβάλλει σε όλε τι χώρες να αυξήσουν τις προστατευόμενες περιοχές τους και να αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί και ε, αναπτύσσεται η οικονομία μας. Πρέπει να πιέσουμε για ένα στόχο 30% για τους θαλάσσιους και χερσαίους πόρους και την προστασία τους. Αυτά όλα επηρεάζουν το σέλος και τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δράσει αμέσως ως μεγάλος ε, πρωταγωνιστής στη συνάντηση, στη συνάντηση του Κονμίν. Με στόχους δεσμευτικούς πρέπει να αποκαταστήσουμε και περιοχές που έχουν καταστραφεί. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα της προστασίας της βιοποικιλότητας και της αναστροφής της διαδικασίας και αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στους στόχους. Επίσης να αναφέρω ένα άλλο θέμα, ε, μια μεγάλη πρόκληση που έχει να κάνει με την ανθρώπινη τεχνολογία, δηλαδή τα γενετικά. Υπάρχουν εταιρείε και οργανισμοί που αναπτύσσουν τεχνολογικές λύσεις οι οποίες μπορούν να εξαλείψουν ολόκληρους πληθυσμούς κουνουπιών, ας πούμε, ε, στην ε, φύση. Και εμεί θέλουμε ένα μορατόριο για τη χρήση τέτοιων τεχνολογιών να μην χρησιμοποιηθούν ε, αφού έχουν συνέπειε τελείω απρόβλεπτες και εντελώ αμετάκλητες. Ευχαριστώ.